todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 um da, da, Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε τη σημερινή μα συνεδρίαση, το σημείο 1 τη σημερινή διάταξη. Το σημείο λοιπόν 1 τη σημερινή διάταξη είναι η έγκριση του σχέδιου ημερησίας διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στις ανακοινώσεις. Ε, έχετε όλες ε, τις ε, γλώσσες διαθέσιμες πλην των μαλτέζικων. Δεύτερο σημείο είναι οι ανακοινώσεις για τους μέρες διαλόγους. Η κυρία Μπλικεβίτσιος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα ε, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην ε, παγκοσμιοποίηση. Πριν από δύο εβδομάδες έγινε ε, ο πρώτος τριμερής διάλογος. Είχε προηγηθεί συνεδρία των σκιωδών εισηγητών όπου συζητήθηκε το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολιτικοί ε, τριμερείς διάλογοι. Και σε αυτή τη συνάντηση είπαμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την άποψη της ηγεσία τελικά του ευρωπαϊκού διαλόγου, ότι δηλαδή ο πολιτικός διάλογος, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν αν δεν ε, έχουμε κάποια βεβαιότητα σε σχέση με το προσεχές πι πι διότι δεν γνωρίζουμε τα ποσά, δεν γνωρίζουμε ε, ποια θα είναι η κατανομή των κονδύλων, άρα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τέτοιου είδους συζητήσει. Για τον πρώτο τριμερή διάλογο, Ε, έγινε η πρώτη συνάντηση, δεν θα συνεχιστεί ε, σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα γίνουν τεχνικές συναντήσεις. Χθε έγινε η πρώτη και κράτησε τρεις ώρες συγκεκριμένα. Είχαμε πολύ έτσι εντατικές συζητήσεις, προσπαθώντας να καταλήξουμε σε συμβιβασμό πάνω σε κάθε ένα από τα σημεία που μας απασχόλησαν. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν σημειώσαμε και σημαντική πρόοδο. Πάντως ε, Υπήρχε πολύ ευνοϊκό κλίμα ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα συνεχίσουμε ε, με τις τεχνικές αυτές ε, συναντήσεις. Επόμενη έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου. Όπως είπα, θα προβλέπονταν και πολιτικοί, πολιτικές διαπραγματεύσεις, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε σήμερα το Σύνοδο Κορυφής που θα συζητήσει το ΠΔΠ. Όμως οι πολιτικές διοργανικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, όσο δεν ξέρουμε τα ποσά. Αυτό είναι απαραίτητο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλω να σας πω επίσης ότι έχω στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησα οι πιο σημαντικές προτάσεις για την συνέχιση του, των προγραμμάτων ε, σε σχέση με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να κατατεθούν νωρίτερα, πριν δηλαδή ε, τα τέλη Δεκεμβρίου ή τις αρχές του έτους, αν δεν έχουμε μέχρι τότε κάποια θετική εξέλιξη. Τα πάντα είναι δυνατά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο και βέβαια θα ακολουθήσουμε τις υποδείξεις της ηγεσία του Κοινοβουλίου. Πενεθήκαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή, όπως είπα, ζητώντας ε, την ε, συνέχιση των προγραμμάτων υπό το Ταμείο για την ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Αυτά και αν υπάρχουν οποιαδήποτε ανώτερα θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε στο σημείο 3 που είναι τα πρακτικά έγκριση των πρακτικών προηγούμενων συνδυάσεων. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Ωραία. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποια παρατήρηση και προχωρούμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, των ε, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Μανουέλ Πιθάρο είναι εισηγητή μας. Είναι στην αίθουσα όμως. Δεν τον βλέπω. Δεν έχει ακόμη καταφθάσει ο Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος σκιώδη εισηγητή που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Εσείς παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο να σας μιλήσω εκ μέρους του εισηγητή που δυστυχώς σήμερα είναι άρρωστος. Αν δείτε τις ε, τροπολογίες βλέπουμε να αναδύεται μια συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για τη συνέχιση αυτού του δικτύου και τα πρώτα χρόνια πρόδευσε το δίκτυο και έχει προσφέρει προσθεμένη αξία στα μέλη. Επίσης έχουμε προσαρμογή στην προεγματικότητα των υπηρεσιών, της απασχόλησης σε σχέση με τις ελευθερίες που παρέχει το πλαίσιο. Φυσικά υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Η, το ΕΛΚ πιστεύει ότι θα πρέπει τα μέλη του δικτύου να τάξουν κάποιες προτεραιότητες ακριβώς όπως έχει πει ο σχεδόν και θα πρέπει επομένως να δούμε το πώς δεν θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα ευρύες διαστάσεις το δίκτυο και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια ακριβώ να δούμε τι θα γίνει τι προτεραιότητε και το ΕΛΚ έχει επισημάνει διάφορα σημεία ότι χρειάζεται κάποιο είδου επαγγελματική κατάρτιση που να αντιστοιχεί στι ανάγκε του επιχειρηματικού κόσμου, ευκαιρίε, ε, και προκλήσει της ψηφιακή τεχνολογία, επίση επίσης προσφορά και ζήτηση στην αγορά απασχόλησης, συνεργασία με επίσης υπηρεσίες απασχόλησης. Και να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο και είμαστε κατά των τροπολογιών των πρασίνων όσον αφορά μία μόνιμη δομή για το δίκτυο. Περιμένουμε τις επόμενες συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, το λόγο έχει ο σκιώδης ή η σκιώδης του Ρινιού, Βέλη. Και εγώ, συναδελφοί, να ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν για αυτές τις θετικές τροπολογίες. Πιστεύω ότι σε πολλά σημεία μπορούμε να τα βρούμε και συμφωνώ 100% ότι θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση υπέρ της απασχόλησης και σταθερότητας των θέσεων εργασίας θα πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η συνεργασία με κοινούς εταίρους όσον αφορά το δίκτυο. Ναι, χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και έτσι να εξασφαλίσουμε ένα στεγανό συνεπές πλαίσιο για να βοηθηθεί η αγορά απασχόληση. Κάτι άλλο σημαντικό για μας είναι να δούμε πώς θα είναι αποτελεσματικέ οι πολιτικές για να βοηθήσουμε διάφορες κοινωνικές ομάδες και κυρίως τους ανθρώπους με αναπηρίε και να δούμε τι θα γίνει με την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, ευκαιρίες που προσθέτει αυτή η τεχνολογία και η ψηφιακή μετάβαση και αλλαγή. Επίσης, να κάνουμε ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, περίοδο διάρκειας του δικτύου. Αυτά να τηρήσουμε. Και τώρα, Στεφανία Ζαμπέλη, για το ID. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που είχε ε, πολύ καλή επίπτωση ε, επί των πολιτών της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το 2027. Είναι σημαντικό βεβαίως να μεταρρυθμιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης γιατί δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες αυτές οι υπηρεσίες σε διάφορες χώρες άρα δεν ε, παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους ε, ε, πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω υποβάλει τροπολογία σχετικά με την ψηφιοποίηση κυρίως. Έτσι θα βελτιωθεί η πρόσφορα διασφαλίζοντας δύο στοιχεία. Πρώτον, καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας και δεύτερον, τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Επίσης, θεωρώ θεμελιώδου σημασία την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών, έτσι ώστε ε, οι πιο, τα πιο προχωρημένα κράτη να βοηθήσουν αυτά που ακόμα βρίσκονται στην πορεία. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι η το δίκτυο ε, των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης ε, ε, μπορεί να αποτελέσει κάτι παραπάνω, χωρίς όμως να περιορίζει τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Σαντορή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Σαντορή από τους πράσινους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή τη συλλογική εργασία επί του θέματος αυτού. Θέμα το οποίο στην αρχή μπορεί να φαινόταν τεχνικής φύσεως, ωστόσο είναι πρωταρχική σημασία για τους πολίτες μας. Πιστεύω ότι ο συντονισμός των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ε, κοινής χρήσης ε, στοιχείων. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες σχετικά με την οικολογική μετάβαση γιατί η ε, μετάβαση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει καλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης στους πολίτες μας καθώς επίσης ε, και για θέματα όπως είναι η πιο προσωπική και εξατομικευμένη παρακολούθηση των ανέργων. Χαίρομαι γιατί έχουν δεσμευτεί όλες οι ομάδες και νομίζω ότι έχουμε περίπου 60 τροπολογίες ε, στο σύνολο και οπωσδήποτε η συζήτηση μεταξύ μας θα επιτρέψει στον εισηγητή κύριο Πιθάρο να ε, προχωρήσει σε καλές συμβιβαστικέ. Ε, χαίρομαι που γίνεται συζήτηση για αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Τα σύμβολα είναι πολύ σημαντικά εις την πολιτική ο ιδιωτικό τομέα οργανώνεται μόνο του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, θεωρώ ότι και ο δημόσιος τομέα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να οργανωθεί αντιστοίχω. Βεβαίω, θα έχετε καταλάβει ότι μέσω της τροπολογία μας δεν δίνουμε λευκή επιταγή στις κυβερνήσεις αλλά πραγματικά θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα, ένα, να περάσουμε ένα σύμβολο βιωσιμότητας ε, και βεβαίως με χαρά θα συμμετάσχω στις συζητήσεις που θα έχουμε με τον κύριο Πιθάρο, τον εισηγητή και τους συναδέλφους συντρόφους, ε, συγγνώμη, σκιώδεις εισηγητέ έτσι ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. το ECR. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, διάβασα τις ε, τροπολογίες και έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Κυρίως ε, όσον αφορά το πρώτο τμήμα κατά κάποιες απόψεις οι τροπολογίες οι οποίες ασχολούνται με αρμοδιότητες ασχολούνται με αρμοδιότητε ε, που είναι όμω αποκλειστικέ αρμοδιότητε των κρατών μελών όπω είναι η κατάρτιση ή ε, όπως η επαγγελματική καθοδήγηση. Επίσης γίνεται λόγος για υγεία, για τη νέα πράσινη συμφωνία. Αυτά εκφεύγουν του πλαισίου. kierunku działań χρειαζόμαστε χρόνο έτσι ώστε να αξιολογήσουμε ε, την σημασία αυτών των δικτύων. Ε, ναι, είναι γεγονός ότι μπορούμε να συζητήσουμε για την Πράσινη Συμφωνία γιατί φαντάζομαι ότι αποτελεί προτεραιότητα ε, και για την αγορά εργασίας αλλά δεν είναι ε, η μοναδική, το μοναδικό πεδίο στο οποίο μπορεί να, να παίξει ας πούμε αυτό το θέμα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Επίσης, συνεργασία με τρίτες χώρες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επίσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως άλλωστε και η μεταναστευτική πολιτική. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν με ποιον και με ποιο τρόπο επιθυμούν να συνεργαστούν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Αρβανίτεκ μέρος της Γκουέντζιελ. Οπότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πιθάρο. Συγγνώμη που αρχίσαμε χωρίς να είστε εδώ, αλλά δεν είχαμε και χρόνο. Παρακαλώ. Έχετε εσείς τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, γιατί άργησα. Αγαπητοί συντρόφοι και θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αυτή η έκθεση. Έχω λάβει 59 τροπολογίες, πολλές από τις οποίες πιστεύω θα βελτιώσουν το περιεχόμενο της έκθεσης και πολλές, ακόμη και αυτές με τις οποίες δεν συμφωνώ, νομίζω ότι θα μας επιτρέψουν να εμβαθύνουμε τον πολιτικό διάλογο πάνω στο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να καταθέσω και εγώ τροπολογίες που θα μας βοηθήσουν να επικαιροποιήσουμε τις προτάσεις μας για αυτό το δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πραγματικότητες. Θέλω να δοθεί σημασία στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και στην ισότητα των φύλων. Είναι ένα θέμα που Νομίζω πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία, όπως ε, επίσης και στους ε, μακροχρόνια ανέργους ε, ή σε άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι να γίνει μία στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Κάτι που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι και οι στόχοι των δυτικών συνθήκων της Ένωσης σε σχέση με την απασχόληση, την κοινωνική πρόοδο ή ε, τον εκάρσιο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να εξυγχρονιστούν αυτές οι υπηρεσίες απασχόλησης γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που ανακύπτουν στην αγορά εργασίας και που οφείλονται και στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις διάφορες αλλαγές που προκαλούν αυτές στις αγορές εργασίας. Και νομίζω ότι πολλές από τις τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση ε, στοχεύουν να συμπεριλάβουμε με διαφορετικές έτσι, αποχρώσεις αυτές τις ε, αναγκαιότητες. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε κάποια πιο λεπτά ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το δίκτυο και το κοινοβούλιο. Υπάρχει μια πρόταση το κοινοβούλιο κάθε 7 χρόνια να λαμβάνει απόφαση και μια δεύτερη άποψη που τη σέβομαι αλλά δεν συμφωνώ είναι ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο να δημιουργήσει ε, ένα δίκτυο που θα λειτουργεί μόνιμα και απλά να κάνει κάποιες αξιολογήσεις ε, καιρούς καιρών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχει νομοθετικό ρόλο και ενεργό μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην είναι απλά παθητικός ο ρόλος του, δηλαδή να γνωμοδοτεί πολύ απλά ε, νίωτε. Νομίζω ότι οι στόχοι που ανέφερα θα επιτευχθούν καλύτερα αν διατηρηθεί ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου. Ένα άλλο σημείο που δημιουργεί έτσι επίσης κάποιες αντιπαραθέσεις ε, και αποκλήσεις απόψεων είναι τι γίνεται με τις τρίτες χώρες και τη συνεργασία τους με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. 31 ε, Δεκεμβρίου οριστικά θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι τρίτη χώρα. Και ε, εκεί ε, ζητήματα που πρέπει, ζητήματα που πρέπει να δούμε. Υπάρχουν επίσης δημοσιονομικοί περιορισμοί του δικτύου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία. Θα πρέπει να γίνει από κάποιο διαφορετικό πρίσμα. Έχει πάντως ε, προστιθέμενη αξία και εγώ θα προσπαθήσω γενικώ να συντάξω μια έκθεση ισορροπημένη που να λαμβάνει υπόψη την πλειοψηφία των βουλευτών τη επιτροπή Μα Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροντινέλη, τους είμαι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών της απασχόλησης μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ καλό στοιχείο όσον αφορά την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Άρα συμφωνώ με τον εισηγητή που υπογραμμίζει αυτή την προσέγγιση. Έχω υποβάλει τροπολογίες ε, ε, σχετικά με δύο θέματα σημαντικά κατά την άποψή μου σε αυτήν την ευαίσθητη φάση χρειάζεται ενίσχυση της συνεργατικής εργασίας ε, του, του δικτύου δημοσίων υπηρεσιών. Να μην είναι αυτός σκοπός, αλλά λειτουργικό στοιχείο με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ε, η πράσινη συμφωνία για την οποία όλοι πρέπει να συμβάλλουν. Η, ε, η πράσινη συμφωνία σημαίνει για να εφαρμοστεί ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μεταβατικό μοντέλο, αλλά κυρίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια σωστή και δίκαιη για όλους μετάβαση που θα επιτρέψει σε όλους να μεταρρυθμιστούν χωρίς όμως να χαθούν θέσεις απασχόλησης. Ε, είσαστε πάρα, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούν να ακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη πάντοτε με αγχώνει ο κόσμο, ο χρόνος που περνάει και δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου, ενάμιση κλπ. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι εάν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, οπωσδήποτε θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος στους πολίτες και επομένως εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε ε, παίξει τον ρόλο μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την εισηγήτρια και όλους τους σκιώδης εισηγητές. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Πάρα πολύ σωστή δουλειά από όλες τις πλευρές και θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι λαμβάνεται υπόψη το ότι το δίκτυο είναι ένα μέσο υποστήριξης του έργου των ε, κρατικών υπηρεσιών απασχόλησης των μελών. Δεν προεδρεύουμε εμείς στο δίκτυο, αλλά αυτές οι εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης πρόκειται για ένα μέσο πολιτικής που βοηθάει αυτές τις υπηρεσίες για το σπουδαίο τους έργο υλοποίησης της πολιτικής που το Κοινοβούλιο ως ε, νομοθέτης θεσπίζει όπως την εγγύηση για τη ε, νεολαία, την ε, πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οπότε συνεχώς υπάρχει εξέλιξη και αναβάθμιση του δικτύου. Απλώς ως σχόλια έχω να πω ότι είναι πολύ θετικό το μήνυμα για την ψηφιακή τεχνολογία και για το ότι θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στην Πράσινη Συμφωνία ε, και οι άλλες ε, τροπολογίες είναι θετικές. Όλες οι προτάσεις δηλαδή που διατυπώνονται μέσα από αυτές τις τροπολογίες. Τώρα όσον αφορά την ε, παράταση της ζωής του δικτύου, γενικά το χρονικό πλαίσιο είναι θέμα προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει πρόθεση του να σταματήσει η λειτουργία του δικτύου, αλλά όπως αναφέρεται μπορούν οι συνομοθέτες να παρέμβουν ε, και να ενημερώσουν, να επικαιροποιήσουν το δίκτυο. Υπάρχει διεθνή συνεργασία, ε, το προβλέπει η απόφαση. Αλλά να μην το παρακάνουμε, μην δίνουμε ε, υπερβολική έμφαση στον διεθνή χαρακτήρα. Σας ευχαριστούμε για όσα κάνατε και για την υποστήριξη σας. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, θέλει τίποτε να προσθέσει ο εισηγητής ή οι σας επενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. 30 Ιανουαρίου για τις ε, τροπολογίες. Ε, συζητήθηκε σήμερα 20 του μηνός και πρόκειται να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας 26 Τρίτου. Και τώρα πάμε στις ψηφοφορίες ηλεκτρονικά. Το πρώτο. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για Συντονισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής όσον αφορά τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης σε σχέση με την έρευνα ανάπτυξης του 20. Α, μισό λεπτό. Queria έχω πρώτα πρώτα μια ανακοίνωση, λέει η πρόεδρος. Έχουμε... Έχουμε θέμα με το Renew. Έχουμε αυτή τη στιγμή 53 μέλη της Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουν 55. Συμβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. α. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν εννέα. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, όχι, εγκρίνεται. Διορθώνει η πρόεδρο. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Εν. Συμβαστική εν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή. Συμβαστική ή e. υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Please repeat um, the compromise we're voting for. When you... Μπορείτε να επαναλάβετε για, για ποια συμβαστική ψηφίζουμε. Πρόκειται για τη συμβαστική Ι, e, ε, λέει ο πρόεδρος. Abrimos a votação. Quem é, contra, quem Ψηφίζουμε τη συμβαστική Ι e και κάνουμε, διορθώνει πρόεδρος, κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. Houve uma Συγγνώμη για τη σύγχυση. Κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το E. Πέρασε ο φορείο. Όχι, όταν ηλεκτρονική δεν χάσταν να λέμε υπέρ κατά, λέει η πρόεδρο. Οπότε απορρίπτεται. Συμβαστική D, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 150, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ε, ε, τι γίνεται, ε, αργεί κάπως να έρθει η μετάφραση από τα πορτογαλικά και γι' αυτό έχουμε κάποιο μπέρδεμα όσον αφορά το τι ψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να τα πω λίγο πιο αργά. 156. Πρώτο τμήμα. Κόντρα. Περ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Compromisso G Συμβαστική G, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική H, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. συντροπολογία τροπολογία 188 ε, ως προσθήκη το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 188. Το δεύτερο τμήμα. Πέρα 188. Απορρίπτεται. J. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Είμαστε στο L, συμβαστική L. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική KA. Κάπα αλφα, Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. M. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπής Πολιτισμού 5. Υπέρ. Όχι. Ξανά από την αρχή λέει ο πρόεδρο. Καλτ, πολιτισμού. πέντε, υπέρ, κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. AQ υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική R, ρο, υπέρ, κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική P. Π, ξαναλέει πρόεδρος, υπέρ, κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων Υπαριθμών. πώ, πώ, όχι, όχι, διόρθωνε πώ Q, Q, συμβαστική Q. Q. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την συμβαστική Q. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και όχι, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά, λέει η πρόεδρο. Εμμέντα 183. Quem vota a 183. Contra? Abstenção. Αποχές. A votação está aberta. Για το 183, κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για το 183. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 127, όχι, διότι καταπίπτει. Yes, false, sim. Emenda 131. Quem vota 131. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική S υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική TAF υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική U. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Β. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 281. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α τάφ υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική X Χ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Y ελληνικό, υπέρ, Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Z. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Τροπολογία 28 ε, ως ε, προσθήκη στη συμβαστική Z. «328 διόρθωσε η πρόεδρος, γιατί είπε κάτι άλλο πριν. Πρόκειται για προσθήκη στη συμβαστική Z, επαναλαμβάνει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 328. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική AC υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 320 τμήμα δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 320 δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτωται. Πρέπει να επαναλάβουμε, λέτε, ρωτάει η πρόεδρος. Ε, Θα κάνουμε επανάληψη ψηφοφορίας. 320. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 338 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 339 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές αναφορές Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2, 4 και 14 είναι ταυτόσιμες, επομένως υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 10 <laughs> συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 πλέον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική AR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG, J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AK, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία επί του τροποποιημένου κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια, την κυρία Ντόμπρεφ και προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία. ό,τι αφορά τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωση για την αναπηρία μετά το 2025 υπέρ, κατά, εποχέ. εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε παρακαλώ την 149. Άρχεται η ψηφοφορία, έχετε ψηφίσει όλοι πέρα ψηφοφορία. Έγινε δεκτή η τροπολογία αυτή. 150 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 6 συμμεβαστικοί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. θα ψηφίσουμε ε, στη, για την τροπολογία 229 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. A favor. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 225 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 233 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Compromisso 8 a favor contra Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δυο τροπολογία 241 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 257. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 275 276, 277 και 278 για αφού πρόκειται για ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα των τροπολογιών 275, 276, 277, 278. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επειδή τα λέτε στα πορτογαλικά, ε, έρχεται μετά από δύο, έρχεται με κάποιο διπλό χρόνο μετάφραση, δύο μεταφράσεις πολλές φορές. Ε, περνάμε από δύο γλώσσες ε, και γι' αυτό αργούμε, καθυστερούμε να ακούσουμε. και υπάρχει και στην περίπτωσή μου ανάγκη να γίνει και διερμηνία στην νοηματική Οπότε καθυστερούμε. Σας παρακαλώ, μπορείτε και εσείς λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. ...286 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 288 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ Ah, Compromisso 18 a 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 305 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβεβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολόγια 298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 326 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 326. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 325 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 338 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 354 υπέρ, 343 ψηφίστηκε μαζί με την προηγούμενη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 310 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 310. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίες Εγκρίνεται 308 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 356 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 360 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, υπέρ, να ξαναρχίσω από την αρχή. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 381 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται θα ελέγξουμε όμως την 381 άρχεται ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας τελικά εγκρίθηκε συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 412 περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 413 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 414 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 416 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 427 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 428 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 4.28 άρχεται η ψηφοφορία αν ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 429 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 430 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 432 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 434 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε τώρα διάφορες τροπολογίες 410, 445, 447, 448, 456. Υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγα λοιπόν ότι ψηφίζουμε μαζί την 410, την 445, την 447, την 448 και την 456. Ψηφίζουμε ομού αυτές τις τροπολόγιες είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ όλων αυτών. Κυρία Γιονκέριος, θα ήθελα να ψηφίσουμε χωριστά την 445. Γιατί έχουμε κάτι άλλο. να είναι ταυτόσιμες, λέει η Πρόεδρος. can go. Συγγνώμη, ε, με ακούλπα. Να προχωρήσουμε. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν όμως, αυτές τις τροπολογίες που είπα, ψήφι Κατά. Αποχές γκρίνονται. Πηγαίνουμε σε 351 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 454 και 462 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 455 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πηγαίνουμε στις αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές Τροπολογία 1 Κατά τι Πάμε στην 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4, 5, 6 από κοινού. Τις ψηφίζουμε ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 9, 28 από κοινού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ καταπίπτει Πού πάμε λοιπόν 26, 27, 42, 51, 52, 53. Μαζί όλες αυτές. Μέχρι και την 64, έτσι, εκεί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα 29, 30, 49, 57, 58 και 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές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 Μάλλον 38, 39 και 40. Όχι, διορθώνει πρώτα. 38 και 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41, 43, 44, 45, 46, 47. Από κοινού όλες αυτές ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 μαζί με 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε ελέγχουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίθηκε 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 90 και η 93 όχι πάμε στην συμβιβαστική 3 λέει πρόεδρος κατά αποχές εγκρίνεται 94 ψήφι Περ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 λέει πρόεδρος συγγνώμη 108 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 Θέλετε να ελέγξουμε την 122, άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι. Απορρίφθηκε. 123 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 125 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την ε, τροπολογία 128 άρχεται η ψηφοφορία σφίσα όλοι πέρας ισοπαλία. Άρα απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλλον ελέγχουμε. Καλύτερα να παληθεύσουμε τα 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Το ίδιο πάλι. Ισοψηφία και πάλι. 26 όλα. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα 134, 137 από κοινού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα, όπως ε, τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 52 ψήφισαν, 52 υπέρ. Συγχαρητήρια. Τώρα πάμε στην τελευταία ψηφορία, λέει η Πρόεδρος, πρόκειται για τις ε, γενικές κατευθυντήριες όσον αφορά την προετοιμασία του προϋπολισμού του 21 τρίτο τμήμα και αρχίζουμε. Πρώτη τροπολογία, υπέρ. Ε, και βάτε κόντρα. Abstenção. Eh, foi Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Ένα. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Λειτουργός έλεγχος για το 10. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι κρίνεται να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 11. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Του 13 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του 13. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 14 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη το αποτέλεσμα, οπότε κάνουμε έλεγχο για το 15. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρασε. Και... Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγραφός 10, 24. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του κειμένου, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται.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 και εμείς